4 του εσωτερικού κανονισμού. Η σειρά των εκλογών είναι η εξής. Πρώτα θα πρέπει να εκλέξουμε πρόεδρο και μετά καθένας από τους τέσσερις αντιπροέδρους διαδοχικά. Πάμε στο σημείο 2 της σας διάταξη, την εκλογή του νέου προέδρου ή της νέας προέδρου. Με ενημέρωσαν ότι οι αναπληρωτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία είναι ο κύριος Φίσας που αντικαθιστά τον κύριο Σφέρ, ο κύριος Βίνκλαρ, που αντικαθεστά τον κύριο Τούτη και ο κύριος Μαραγκάλιο που αντικαθιστά την κυρία Evans. Να επιστήσω την προσοχή των πολιτικών ομάδων στο εξή. Αν συμβεί κάποια αλλαγή πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος πριν να ε, ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ορίστε, κύριε Καστνοντέμσκι. Εκτός μικροφώνου και ο Ανάψτε το μικρόφωνο, λέει η Πρόεδρο. Είμαι τον κύριο Λούις αντικαθιστώ. Είμαι αναπληρωτής του κύριου Λούις. Thank you. Are additional... Υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις, κάποια άλλη πληροφορία. Όχι. Καταρχάς, να διαπιστωθεί ύπαρξη απαρτίας. Οκτώ μέλη, το εντέταρτο των μελών. Δεν υπάρχει πρόβλημα βέβαια, διότι λίγο πολύ όλα τα μέλη είναι παρόντα. Θα ζητήσουμε διορισμό, μάλλον υποψήφιο για τη θέση του Πρόεδρου. Κυρία Καμάη. Προτείνουμε την κυρία Σιλβία Κώστα ως Πρόεδρο της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Μου είπαν ότι η κυρία Σίλβια Κώστα υποψήφιος είναι πλήρες μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού, αντιπροσωπεύει πολιτική ομάδα και έχει συμπληρώσει και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Ρωτώ τώρα την υποψήφια εάν συμφωνεί να υπηρετεί σε αυτή τη θέση. Απάντηση ναι, συμφωνώ, λέει η κυρία Κώστα. Εφόσον υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, προτείνω κυρία Σιλβία Κώστα να εκλεγεί διαβοής. Αγαπητή Σίλβια, συγχαρητήρια και σε καλό να έρθεις να πάρεις την θέση της Προέδρου. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ σύντομα Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω πολύ για την υποστήριξή σας. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να εγγυηθώ να τηρούνται οι κανόνες στη λειτουργία της Επιτροπής και θα, θα αξιοποιήσω και την προσπάθεια όλων σας. Ο πολιτισμός και η παιδεία μαζί με τις πολιτικές για την νεολαία και τις αθλητικές αξίες ε, είναι η βάση για την Ευρώπη για να ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη γραμματεία τους διερμηνείς επίσης για τη δουλειά που κάνουν και θα συνεχίσουμε με την εκλογή των αντιπροέδρων. Λοιπόν, θα συνεχίσω ιταλικά. Αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τους αναπληρωτές, να μας το γνωστοποιήσετε αν έχει αλλάξει κάτι σχέση με την πρώτη ψηφοφορία, όχι. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο κύριος Βίνκλερ αντικαθιστά τον κύριο Τότι, ο κύριος Μαργκάλ αντικαθιστά την κυρία Evans και ο κύριος Φίσας αντικαθιστά τον κύριο Σβέρ και Κραντέσκι αντικαθιστά το συνάδελφο Lever. Έτσι. Καλώς μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει απαρτία, υπάρχει απαρτία. Οπότε ζητώ να μου πείτε ποιοι είναι υποψήφοι για τη θέση πρώτη αντιπροέδρου. Κυρία Βεράιαν. Καταρχάς να σας συγχαρώ για την εκλογή σας εκ μέρους του ΕΛΚ προσδοκούμε να έχουμε μια καλή συνεργασία μαζί σας όπως και στην προηγούμενη θητεία. Ως ε, ΕΛΚ θα ήθελα να προτείνω τον, την κυρία Αντρέα Μπόξκορ για πρώτη αντιπρόεδρα. Ευχαριστώ. Σαμπίν Βεράιαν μας ενημέρωσαν ότι η υποψήφια Ανδρέα Βόξορ είναι μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού υποστηρίχθηκε από πολιτική ομάδα και έχει συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Ζητώ από την υποψήφια αν δέχεται να αναλάβει αυτό το καθήκον της θέσης Αντιπροέδρου. Καλώς. Υπάρχει μόνο μία υποψηφιότητα για θέση Αντιπροέδρου, πρώτη Αντιπροέδρου. Προτείνω η κυρία Αντεμπόξορ να ε, εκλεγεί δια βοής. Σας συγχαίρω βέβαια και σας καλώ να έρθετε εδώ να πάρετε θέση στη θέση του Προεδρείου. Κύριε Μποσχούρ. Eh, mm, Τώρα, εφόσον υπάρχει ίδια παρτία, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ποιο είναι υποψήφιο για θέση δευτέρου αντιπροέδρου. Ορίστε. Ε, Σα ευχαριστώ. Από πλευρά των φιλελευθέρων, προτείνουμε τον κύριο Γιακανό ο οποίος έχει διατελέσει στην ε, Ρουμανία υπουργό Πολιτισμού και θέλουμε θα είναι ο καλύτερος δυνατός υποψήφιος για αυτή τη θέση. Σας ευχαριστώ. Οπότε με ενημέρωσαν ότι υποψήφιος ο κύριος Γιάκονο είναι μέλος Επιτροπής Πολιτισμού. Υπο... Είναι υποψήφιος πολιτικής ομάδας και συμπλήρωσε τη δήλωση όσον αφορά τα οικονομικά της συμφέροντα. Ρωτώ τον κύριο Γιακονού εάν συμφωνεί να αναλάβει αυτή τη θέση. Ορίστε. Μάλιστα, καλώς, έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, οπότε και σε αυτή την περίπτωση προτείνω να εγκριθεί ο διορισμός σε θέση αντιπροέδρου ε, διαβοής, να εγκριθεί η ανάληψη των καθηκών του κύριου Γιάκονου. Και σας παρακαλώ να έρθετε να καθίσετε εδώ στη θέση του Προεδρείου, κύριε Γιακόνο. E, Πάμε λοιπόν στην εκλογή τρίτου αντιπροέδρου. Ποιος είναι υποψήφιος για την θέση αυτή. Ορίστε. Ε, yes, ε, από πλευρά των Πρασίνων, σας προτείνουμε την κυρία Τρούπελ, την κυρία Χέλγα Τρούπελ, σαν τρίτη αντιπρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Τρούπελ, συμφωνείτε. Ναι, συμφωνώ, λέει η κυρία Τρούπελ. Χαίρομαι που συμφωνείτε. Ε, ε, ενώ θα, θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Η υποψήφια είναι η κυρία Χέρκα Τρούπελ, μέλος τη Επιτροπής Πολιτισμού. Την ε, πρώτη είναι πολιτική ομάδα και συμπλήρωσε και τη δήλωση όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα. Κυρία Τρούπελ, παρακαλώ να έρθετε εδώ στη θέση του Προεδρείου συγγνώμη, λέει πρόεδρο, ξέχασα το πιο σημαντικό. Συγγνώμη, συγγνώμη, τουλάχιστον σήμερα. Προτείνω να εκλεγεί διαβοή, λοιπόν. Ε, με προλάβατε δια του χειροκροτήματό σα, αλλά έπρεπε να το πω αυτό. Συγχαρητήρια, λοιπόν, στην κυρία Τρούπελ. A questo punto chiedo la... Υποψήφιο για θέση τέταρτο αντιπροέδρου θα θέλαμε τώρα. Ποιος προτείνει. Ορίστε κύριε Βεράιαν. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προτείνουμε την κυρία Μικαέλα Σόλτροβα. Eh, Καλώς η υποψήφια Μικαέλα Σόλτροβα είναι μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού, προτάθηκε πολιτική ομάδα και συμπλήρωσε τη δήλωσή της περί οικονομικών συμφερόντων. Ρωτώ λοιπόν την κυρία Σόλτοβα αν δέχεται να είναι υποψήφια. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, συγγνώμη. Έχουμε μία μόνο υποψήφια. Προτείνω λοιπόν να εκλέξουμε την κυρία Σόλτοβα δια βοής και την παρακαλώ να έρθει εδώ στις θέσεις του Πρόεδριου. Bene. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η εκλογική διαδικασία. Ας πάμε λοιπόν στα άλλα σημεία της ημερήσιας διάταξης της απογευματινής συνεδριάσεως. Πρώτα απ' όλα στο σημείο 4 έχουμε την βεβαίωση του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος για τις συνεδριάσεις ε, του 2014. Πρέπει λοιπόν να επιβεβαιώσουμε, επικυρώσουμε το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα στα έγγραφά σας θα πρέπει να έχετε ήδη λάβει τις σχετικές πληροφορίες, τον κατάλογο των συνεδριάσεων που ενεκρίθηκαν από την απερχόμενη ε, επιτροπή της προηγούμενης θητείας. Δεν ξέρω αν είχατε το χρόνο να διαβάσετε το πρόγραμμα των συνεδριάσεων και αν μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις πέντε συνεδριάσεις που μας μένουν μέχρι το τέλος του 2014 της Επιτροπής μας. Συμφωνείτε? Σημειώσατε δεν ξέρω αν θέλετε να, επαναλάβετε, να επαναλάβω τις ημερομηνίες, τις ξέρετε πιστεύω. Προχωρούμε λοιπόν στην έγκριση του προγράμματος των συνεδριάσεων μας. Βέβαια η πρόταση των συνεδριάσεων για το 2015 θα παρουσιαστεί στη συνεδρίαση των συντονιστών στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Πέμπτο σημείο, τα διάφορα, κάποιες πληροφορίες η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες 3η 22 Ιουλίου για ανταλλαγή απόψεων για τη γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό του 2015. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων εκείνη την ημέρα και 14 Ιουλίου θα γίνει συνεδρίαση των συντονιστών για να διοριστούν οι συγητές για τον προϋπολογισμό του 2015 και να θετηθεί και το πρόγραμμα ε, της διαδικασίας, το πρόγραμμα, η διαδικασία του προπολογισμού. Ζητήθηκε η πρόταση των συνοδιστών να εγκριθεί μέσω email, ε, λόγω ελλείψης χρόνου μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να εγκριθούν οι προτάσεις των ε, συντονιστών, γιατί δεν έχουμε πολύ χρονικό, μεγάλο χρονικό περιθώριο, να υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Δράτω με τις ευκαιρίες και πιστεύω και εν ονόματι της Προεδρίας, του Προεδρίου σας να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε μέχρι τώρα και τη δουλειά που θα κάνουμε μαζί από εδώ και μπρο, μαζί με τη γραμματεία, θα ευχαριστώ τη γραμματεία ε, της Επιτροπής, τους διερμηνείς, τους κλητήρες. Ευχαριστώ όλους και εύχομαι καλή αρχή της νέας θητείας σε όλους σας. Ευχαριστώ. Ορίστε. Κάποιος ζήτησε το λόγο. Κέζος. Έχετε το λόγο. Κύριε Γλέζο, έχετε το λόγο. Το, μικρό, το μικρόφωνο σας παρακαλώ κύριε Γλέζο. Θα ευχηθώ καταρχήν καλή επιτυχία στο έργο του Προεδρείου. Ε, ψήφισα με μεγάλη εμπιστοσύνη και ιδιαίτερα επειδή βλέπω τέσσερις γυναίκες και έναν άντρα. Ελπίζω να μην τον καταπιέσετε αρκετά και να μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του. Θα ήθελα όμως, επειδή διατέλεσα πριν 30 χρόνια μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να γνωρίζω ποιες είναι οι δικαιοδοσίες και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής. Κανονικά. Θα έπρεπε πρώτα από αυτό να αρχίσουμε. Κανονικά, δημοκρατικά. Πρώτα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες μας. Ποιο είναι το περιεχόμενο της δουλειάς μας και μετά να προβούμε στις Αλλά δεν πειράζει. Τώρα μπορώ να μάθω και πιστεύω ότι θα γνωρίζετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες γιατί μαθαίνω πράγματα που δεν υπήρχαν παλιότερα. Παλιότερα είχαμε μεγάλη αυτονομία η κάθε επιτροπή. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό, ναι ή όχι. Λοιπόν, ε, πιστεύω ότι εσείς ε, γνωρίζετε το θέμα και θα ήθελα έναν πρώτο κατατοπισμό γύρω από το πρόβλημα αυτό ποιες είναι οι αρμοδιότητές μας <clears throat> ποια είναι η αυτονομία μας σε σχέση και με την Κομισιόν αλλά και σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με, την, με το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρακαλώ Αξιότιμε κύριε Βουλευτά, μπορώ να απαντήσω εν μέρη γιατί ζητώ συγγνώμη ότι έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας και δεν μπορώ να το αναλύσω όλο. Πρέπει να έρθει εδώ να συνεδριάσει μια άλλη επιτροπή. Να σας διαβεβαιώσω για δύο πράγματα πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα σίγουρα το Προεδρείο θα εγγυηθεί σίγουρα την ισορροπία. Ε, λοιπόν, λοιπόν, δεν θα επικρατήσουν οι γυναίκες δεν θα κάνουμε το λάθος που έκαναν ιστορικά οι άντρες. Σας διαβεβαιώνω, δεν καταπιέσουμε τον άντρα δηλαδή. Για το δεύτερο σημείο που είναι πολύ κρίσιμο σημείο, νομικό και πολιτικό, και αυτό δεν μας διαφεύγει βεβαίως ούτε από εσά. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία για να τα συζητήσουμε, να μπούμε σε βάθος στην επόμενη συνεδρίαση 22 Ιουλίου. Αυτό που θέλω να σας πω, διότι έλαβα και την ευφυή πρόκληση που μου απευθύνατε στην παρέμβασή σας, θέλω να πω σίγουρα αυτή την περίοδο έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητες, έδωσε η συνθήκη της περισσότερες αρμοδιότητες ε, στο κοινοβούλιο σας συνομοθέτη και ε, έναντι των μορφών συνεργασίας που υπάρχουν πάνω τα θέματα για την παιδεία, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό που είναι νέα αρμοδιότητα, για τις πολιτικές για τους νέους και για τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι επιγραμματικά σας τα αναφέρω. Αλλά σίγουρα θα εμβαθύνουμε όπως είναι και σωστό να γίνει και οι συνάδελφοι θα επιθυμούν να γίνει εμβάθυνση, διότι είναι σωστό να ξεκινήσουμε με το γνωρίζοντας ακριβώς ποια είναι η περίμετρος των αρμοδιοτήτων μας. Και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για την καλοσύνη με την οποία παρουσιάσατε αυτά απέναντί σας και τα καλά σας λόγια. Εδώ λοιπόν, κλείνουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ και καλή δουλειά σε όλους.